Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω και αύριο θα δούμε ποιος δηλώνει τι, ποιος πρεσβεύει τι σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λούλινγκ, έχει ολοκληρωθεί ως εκ τούτου η συζήτηση στο θέμα αυτό και αύριο στο 12 μεσημέρι θα γίνουν οι ψηφοφορίες. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη έχει προβλέπει την έκθεση της κυρίας Χούμπνερ σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν επιλούνται από σοβαρέ δυσκολίε όσον αφορά τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Και ξεκινώντα την συζήτηση, θα ήθελα να σα επισημάνω ότι θα είμαι πάρα πολύ αυστηρό προ την τήρηση του χρόνου γιατί έχουμε μόνο μέχρι τι 9 το βράδυ χρόνο δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε περισσότερο τη συνεδρίαση. Το λόγο έχει η κυρία Χιούμνερ για 4 λεπτά η συγγήτρια. Uh, thank you very much. Πρόεδρε, Κύριε Πίτροπε, ευχαριστώ. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια αρχίζω τις δηλώσεις μου εδώ με τη δηλώση ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη στην Ευρώπη και θα το ξαναπώ και σήμερα. Η λιτότητα στις χώρες που πλήττει η κρίση δεν οδήγησαν σε ανάπτυξη λόγω των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα και της έλλειψης ρευστότητας. Χρειάζονται λοιπόν περισσότερε εγγυήσει για να δώσουμε τη δυνατότητα ο ιδιωτικό τομέα να ενεργοποιηθεί περισσότερο σε υλοποίηση έργων, ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κινητοποιήσουμε όλου του διαθέσιμου πόρου για να πρημοδοτήσουμε την ανάπτυξη με ειδικά μέτρα. Και η νομοθετική αυτή πρόταση σε αυτό αφορά. Πρόκειται για ένα εργαλείο επιμερισμού κινδύνου με στόχο να διευκολύνουμε την απορρόφηση των πόρων του Τμήματο Συνοχή και του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτημένων προγραμμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι συγκεκριμένε χώρε. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, καταρχά, έχουμε έργα υποδομών προτεραιότητα, των οποίων η υλοποίηση έχει σταματήσει λόγω ακριβώ τη έλλειψη ιδρυτική χρηματοδότηση. Αυτό αφορά τι μεταφορέ αλλά και περιβαλλοντικέ υποδομέ που μάλιστα αποφέρουν έσοδα και όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορεί να καλυφθεί το κόστος της χρηματοδότησης αυτών των έργων λόγου και των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να μην υλοποιηθούν τα έργα αυτά, διότι, παραλαμβάνω, οι ιδιώτε επενδυτέ και οι τράπεζε είτε δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα για να δώσουν δάνεια, είτε δεν ε, είναι πρόθυμοι πλέον να αναλάβουν τον σχετικό κίνδυνο. Το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπει επίση την δυνατότητα χρηματοδότηση και άλλων έργων τα οποία δεν είναι συγχρηματοδοτούμενα από την συνοχή αλλά τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τη πολιτική συνοχή και που αποφέρουν επιπλέον και προστιμένη αξία στην ευρωπαϊκή πολιτική για ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Το προτινόμενο μέτρο θα υλοποιηθεί από την Κομισιόν βάσει του ενδιαφερμένου κρατου μέλους με την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Τραπεζής Επενδύσεων και σε συνεργασία με ιδιώτες χρηματοδότες. Τα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται θα υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Κομισιόν δηλώνοντα το έργο και την απαιτούμενη χρηματοδότηση, που θα καλύπτεται δηλαδή από το σχετικό μέτρο. Η Κομισιόν θα σταθμίζει την αναγκαιότητα και από εκεί και πέρα θα ενεργοποιεί το μέτρο σε συνεργασία με την ΕΤΕΠ. Ο κανονισμός προβλέπει λεπτομερή περιγραφή της σχετική διαδικασίας για να υλοποιηθεί ο σχετικό επιμερισμό κινδύνου. Επίση, προσδιορίζει το ανώτερο όριο προπολισμού του νέου μέτρου και την αντιμετώπιση των κινδύνων και εκτάκτων περιστάσεων όπως απολειών, ζημιών. Η Κομισιόν θα φροντίσει μόνο έργα τα οποία ικανοποιούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τα οποία έχουν από την ΕΤΕΠ ή άλλο παρόμοιο οργανισμό να επωφελούνται του μηχανισμού. Ελπίζω ότι η ευριανή ψηφοφορία θα επιτρέψει στη συνέχεια και στο Συμβούλιο να εγκρίνει τον κανονισμό ώστε τον Μάιο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δημοσιευθεί το μέτρο στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί βεβαίω. σε ισχύ την ίδια ακριβώς ημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Και τώρα το, νόμο, το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής, ο κύριος Σεμέτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον Ιούνιο του 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθάρρυνε την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προχωρήσουν συνέργειες μεταξύ των ε, προγραμμάτων ε, που υπάρχουν για την Ελλάδα με συνδυασμό των ε, ε, κοινοτικών κονδυλίων. Θα έπρεπε να ενισχυθεί η ικανότητα απορρόφηση των κονδυλίων αυτών και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία ε, ε, ε, θέσεων εργασία. Το αργότερο το 2011 τα κράτη-μέλη ε, της Ευρωζώνης διεύρυναν την εντολή αυτή και κάλεσαν την Κομισιόν και την ΕΤΕ να ενισχύσουν τις ενέργειες μεταξύ των δανειακών προγραμμάτων και των κοινοτικών κονδυλιών σε όλα τα κράτη-μέλη που δέχονται κοινοτική ή διεθνή ε, χρηματική βοήθεια. Τον Ιανουάριο του 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Κομισιόν ε, ε, και την Τράπεζα να ενισχύσουν τις δράσεις αυτές για την υποστήριξη της μεγέθυνσης περιλαμβάνοντας και τη δυνατότητα της χρήσης του κοινοτικού προϋπολογισμού για μόχλευση. Τον Οκτώβριο του 2011 η Κομισιόν ε, υιοθέτησε μια πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου του 2006 1083. Ε, ο σκοπός ήταν να υπάρχει δυνατότητα ε, χρηματοδοτήσεων που έχουν εγκριθεί σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχή και τα Διαρθρωτικά Ταμεία για να δημιουργηθούν ε, εγγύσει και δάνεια ε, που θα δίνονται από την ΕΤΕΚ ή άλλου ε, εθνικού ή διεθνεί οργανισμού με εντολή δημόσιου οργανισμού μέσα από ένα λεγόμενο μέσο επιμερισμού του κινδύνου. Ο στόχο είναι τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρέ δυσκολίε όσον αφορά την χρηματοπιστωτική ε, σταθερότητα και στα οποία έχει δοθεί ε, η οικονομική βοήθεια σύμφωνα με έναν από τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Ο σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά ε, εμπόδια που αντιμετωπίζουν διάφορα κρατημέλη, ιδιαίτερα η Ελλάδα, όσον αφορά την εξέβρεση της απαραίτητης ιδιωτικής ε, χρηματοδότησης για την υλοποίηση διαφόρων έργων υποδομών και παραγωγικών έργων που μπορούν, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από τα δημόσια κονδύλια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για έργα υποδομών που δημιουργούν καθαρά έσοδα. Ε, και η αξία των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από ε, επιδοτήσεις μέσω των μέσων συνοχής. Ε, επίσης, αυτό ισχύει και για την προστασία επενδύσεων, όπου περιορίζεται η κρατική χρηματοδότηση λόγω των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι, θα δοθεί μια απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κρίση. Αυτό όμως δεν αρκεί, ιδιαίτερα για τα έργα που δημιουργούν έσοδα, διότι το κόστος επένδυσης που καλύπτεται από τα έσοδα αυτά δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέτρο που προτείνεται είναι μια εξαίρεση από το συνήθες πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής συνοχής και αιτιολογείται από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλει η κρίση. Ε, από την δημοσίευση της πρώτης αυτής της Κομισιόν ε, μεσολάβησε έντονος διάλογος με το ε, Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής και ιδιαίτερα την κυρία Χιούμπνερ, την πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, για την υποστήριξή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και να ευχαριστήσω τους εισηγητές τους για την υποστήριξή τους. Η έγκριση αύριο της έκθεσης Χιούμπνερ θα ανοίξει το δρόμο για να εξασφαλιστούν ε, στρατηγική σημασία έργα που χρηματοδοτούνται από την πολιτική συνοχή χωρίς να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός που έχει ε, οριστεί για αυτά και ε, με τον τρόπο αυτό θα επανέρχονται κάποιες συνεισφορές στον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό. Ε, θα ε, έτσι, θα διευκολυνθεί η υλοποίηση έργων υποδομών και περιβαλλοντικών έργων, καθώς επίσης και άλλων έργων που είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την Ελλάδα, για την ανάκαμψη και τη δημιουργία εργασίας η υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών και μόνο στον τομέα των μεταφορών ε, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μόνο θα δημιουργήσει 50.000 ε, θέσεις ε, εργασίας. Και άλλα κράτη-μέλη που πλήττονται από την κρίση μπορούν να υποφεληθούν από το προτινόμενο μέτρο. Πέρυσι η πολιτική συνοχή χρησιμοποιήθηκε πολλέ φορέ για να αντιμετωπίσει τι μεταβαλλόμενε ανάγκε ε, των κρατών μελών υπό τι συνθήκε τη κρίση. Ε, μια εξαιρετική διοργανική συνεργασία ε, βοήθησε να δοθεί η ενίσχυση αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καλό λοιπόν του ευρωβουλευτέ να υποστηρίξουν αυτή την νομοθετική πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά κύριε Επίτροπε. Και τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Ριβελίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρόταση τροποποίηση του κανονισμού 1083 του 2006 μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να μεταφερθεί η άμεση, σε άμεση διαχείριση της Κομισιόν ε, κονδύλια τα οποία έχουν ε, ε, προσδιοριστεί για, μέρος, για ενίσχυση των κρατών μελών που κινδυνεύουν να χαθούν λόγω της αδυναμίας υλοποίησης διαφόρων έργων. Η... Εγώ ως της, της Επιτροπής Κοντ θεωρώ ότι το μέτρο αυτό θα είναι στρατηγικής σημασίας για χώρες όπως η Ιταλία που αν και δεν είναι στην ίδια κατάσταση όσον αφορά το χρέος με την Ελλάδα ή την Πορτογαλία πρέπει και αυτή να αντιμετωπίσει την κρίση. Το ζήτημα είναι σαφές. Ε, αν δεν... Ε, ε ο προγραμματισμός που υπάρχει δεν επιτρέπει να επιτευχθούν οι επιδεκόμενοι στόχοι. Η δυνατότητα λοιπόν θα ήταν ε, όχι μια απώλεια πόρων, αλλά ε, μια κίνηση που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να οργανώσουν καλύτερα ε, τις δαπάνες τους σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Η κρίση αυτή η χρηματοοικονομική δεν ε, έχει ε, λυπηθεί καμία από τις χώρες. Άρα το να περιοριστεί σε μία μόνο χώρα ε, αυτό το μέτρο ή σε ορισμένες χώρες θα ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ευχαριστώ για μισή λεπτό τώρα ο κύριος Παπαστάκος, εκμέλους του ΕΛΚ. Αξιολογώς απόλυτα θετική την πρόταση για τη δημιουργία του χρηματοδοτικού μέσου επιμερισμού του κινδύνου με στόχο τη στήριξη έργων υποδομών και παραγωγικών επενδύσεων όπως ανέφερε και η συγγήτρια η κυρία Χιούμπνα πράγματι καθίσταται επιτακτική ανάγκη δημιουργίας συνθηκών οικονομικής μεγέθυνσης σε μια κρίσιμη συγκυρία σε μια οικονομική μετεωρολογία όπου οι δημοσιονομικές περικοπές θίγουν σημαντικά και τις ελληνικές δημόσιες επενδύσεις ενώ η έλλειψη ρευστότητας και πρόσβαση σε χρηματοδότηση δυσχεραίνουν εξίσου και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θέλω να σα πω κυρίε και κύριοι συνάδελφοι ότι κρίσιμα μεγέθη τη ελληνική οικονομία έχουν επιδεινωθεί δραματικά παρά τι πρωτοφανεί θυσίε τη ελληνική κοινωνία. αναφέρομαι πρωτίστω στην εκτόξευση του ποσοστού ανεργία το οποίο αγγίζει πλέον το 50% σε ό,τι αφορά του νέου. Ευελπιστώ ότι τόσο η Κομισιόν όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διασφαλίσουν του όρου, παραδείγματο χάρη ω προ το δίκτυο μόχλευση, και ω προ τι επιλέξιμε επενδύσει για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εν λόγω χρηματοδοτικού εργαλείου με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την πραγματική οικονομία. Τέλο, πέραν τη επιβλημένη δημοσιονομική εξυγίανση, απαιτείται κατά τη γνώμη μου κατεπηγόντως τονίζω κατεπηγόντω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημιουργική αναπτυξιακή φυγή προ τα εμπρό και έξοδο από το φαύλο κύκλο λιτότητα ύφεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Κλέβα, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η εκτέλεση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ερωτικό Ταμείο ε, καλούν ε, για συγχρηματοδότηση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τα κράτη τα οποία έχουν περισσότερο πληγή από την κρίση και λόγω της επιδείνωσης της ε, πιστοληπτικής τους αξιολόγησης δεν μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα. Και έτσι απαιτείται μια εξαίρεση από τον συνήθι ε, κανονισμό για την ε, χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προξενεί η κρίση. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να καλύψει αυτή την διαφορά, αυτό τον κίνδυνο, τον επιπλέον κίνδυνο. Διαφυλάσσονται έτσι και ιδιωτικέ επενδύσει και υλοποιείται ο στόχο της πολιτική συνοχής. Εγκρίνονται κονδύλια που εξυπηρετούν την ανάπτυξη περιφερειών και κρατών και ω εκ τούτου δεν επιβαρύνεται επιπλέον ο προϋπολογισμός των κρατών. Τα μέτρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να οδηγούν στην διασφάλιση της υλοποίησης των έργων εκείνων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τέτοια ε, κονδύλια. Ιδιαίτερα η Ελλάδα έχει ε, μεγάλη ανάγκη από αυτή την στήριξη, περιμένει με αδμονία το πράσινο φως και τα μέτρα αυτά πιστεύω θα αποβούν ει όφελο σημαντικό εκείνων των κρατών που έχουν περισσότερο πληγεί από την κρίση. Χρειάζεται ταχύτατη υλοποίησή τους, ε, γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει θέση σε αυτή τη σημαντική ε, στιγμή και την ανάγκη που αισθάνονται αυτά κράτη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο, εκ μέρου των ε, φιλελευθέρων, η κυρία Μανέσκου. Πρόεδρε, κάθε τροποποίηση κανονισμού με γνώμονα την υλοποίηση προγραμμάτων συνοχής θα έχει θετικό αντίκτυπο στις πληττωμένες οικονομίες. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να εγκρίνουμε αύριο τη σχετική έκθεση όσον αφορά τον επιμερισμό του κινδύνου για τα κράτη-μέλη βεβαίως τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρότερε δυσκολίε όσον αφορά την χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στα κράτη αυτά να συνεχίσουν την υλοποίηση των έργων στον δρόμο τη ανάπτυξη. Πρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει τον σχετικό κανονισμό το συντομότερο δυνατόν. Η ομάδα μας, η Άλτε, υποστηρίζει λοιπόν τον υφιστάμενο συμβασμό, διότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα που εντοπίσαμε. Η ΕΤΕΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των επιλεξίμων έργων. Το νέο μέτρο λοιπόν το υποστηρίζουμε, θέλουμε όμως να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρηματοδοτήσουμε έργα τα οποία δεν είναι οικονομικώς βιώσιμα. Έχει μεγάλη σημασία τα χρηματοδοτούμενα έργα πρώτα να αναλυθούν με βάση μελέτες κόστους ωφέλειας με τρόπο ενδελεχή και με γνώμονα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Και τώρα εκ μέρου ε, της ομάδας των Πρασίνων για ένα λεπτό, η κυρία Σρόντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. το μέσο επιμερισμού του κινδύνου προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευπρόσδεκτο για εμάς πρασίνους. Ως προς την ε, δημοσιονομική τεχνική του ε, αντισυχεί αντιστοιχεί σε μια πράσινη πρόταση για τα broadships και πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε τον ε, δρόμο αυτόν που θα διευκολύνει και την Ελλάδα να βγει από την κρίση. Χρειάζεται λοιπόν να εγκριθεί αυτό το χρηματοπιστωτικό μέσο. Πλην όμως η τροποποίηση στον κανονισμό γίνεται κατά τρόπο ο οποίος δεν εγγυάται κατ' ουδέναν τρόπο την ε, ποιοτική ε, υλοποίηση αυτών των επενδύσεων. Ούτε δηλαδή για βιώσιμη ανάπτυξη ε, μιλάει, ούτε για, ούτε για σταθεροποίηση των θέσεων εργασίας. Επιπλέον αναφέρεται ότι θα πρέπει ε, να οικοδομούνται περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι χάρη στον κανονισμό αυτών. Αυτή είναι σφαλμένη επιλογή. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι επενδύσεις των πολιτών θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε οι επενδύσεις αυτές να είναι βιώσιμες και γι' αυτό δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της ομάδας ε, ECR ο κύριος Φλάσακ έχει το λόγο. Dámy a dnes opatření, se Evropská komise snaží řešit dopady vysokého zadlužení. Κυρίε και κύριοι, εδώ με για μέτρα να βοηθήσουμε κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση στι ιδρυτικέ αγορέ. Για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι βεβαίω ε, πολύ σημαντικό να διευκολύνουμε ακριβώ τι επιχειρήσει να εξασφαλίσουν δάνεια είτε από την ΕΤΕΠ είτε από κάποιον άλλον οργανισμό. Όμω α μην υπερβάλλουμε. Κάθε τράπεζα και κάθε επενδυτική τράπεζα σταθμίζει τους κινδύνους ενός δανείου και καθορίζει ένα επιτόκιο συναφώς. Ο ετών, λοιπόν, λαμβάνει ένα δάνειο με βάση αυτό αλλά και βάση εξωτερικών εγγύσεων. Αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό. Φοβούμαι ότι αν δεν προχωρήσουμε θα συσσωρευτεί περισσότερο χρέο. Καλό λοιπόν όλους να συμβάλλουμε στην βελτίωση της απόδοσης των πολιτικών μας και όχι μόνο να αυξήσουμε τα ποσοστά απορρόφηση. Ευχαριστώ. Εκ ομάδας ε, EFT, ο κύριος Μπάφτον παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η δημιουργία ενό μέσου επιμερισμού του κινδύνου για να διευκολύνει την απορρόφηση ε, των κονδυλίων από ιδιωτική χρηματοδότηση. Αυτός καθεαυτός δεν είναι κακή ιδέα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να εξασφαλίσει ε, το δανεισμό από τον ιδιωτικό τομέα και άρα αποδεικνύει με πόση ε, την αποτυχία των ε, μέσων που έχουν επιλεγεί για την αντιμετώπιση της κρίσης των ευρωπαϊκών κρατών, των κρατών του ευρώ. Ε, προσπαθεί δηλαδή να βρει μικρά όπλα, μικρούς βεληνικούς για να κερδίσει μια μικρή μάχη ενώ ακόμα μένεται ο πόλεμος και δεν έχει ακόμη κρυθεί. Η ευρωπαϊστική αυτή ιδεολογία καταστέλει την ανάπτυξη. Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη. Περιφερειακές, ε, περιφερειακή λοιπόν ανάπτυξη μπορεί να εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα κρατών μελών, αλλά όχι απαραίτητα και επιπλέον αυτό οδηγεί σε μια απόλυτη άρνηση της πραγματικότητας, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι το ευρωπαϊκό ιδεώδες είναι ε, μια αρχή περάνω πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά ο κύριος Στάτλερ έχει το λόγο, τους μη εγγεγραμμένους. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Με τον κανονισμό αυτό η πολιτική συνοχή καθίσταται ε, οριστικά τμήμα της, ε, του μέσω διάσωση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο απορρίπτουμε. Προτείνεται αυτό ω κομμάτι της περιφερειακή ε, της πολιτικής ε, συνοχής λοιπόν. Η κυρία Χιούμπνερ προσπάθησε να μας εξηγήσει τα μέτρα, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η εσωτερική συγκυρία στην Ελλάδα ύστερα από τη διά, τα μέτρα διάσωση, έχει μάλλον επιδεινωθεί και πολύ σημαντικά επιδεινωθεί και βαίνει σιγά σιγά η Ελλάδα προς την ε, πτώχευση με τα μέτρα αυτά. Εδώ γίνεται λόγο λοιπόν στην πρόταση του κανονισμού για μέτρα επιμερισμού του κινδύνου για κράτη τα οποία κινδυνεύουν ή βρίσκονται σε ιδιαίτερε δυσκολίε όσον αφορά την χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Μα οποιοδήποτε έχει συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια ή έχει ε, συνεγγυηθεί βρίσκεται σε κίνδυνο. Εδώ μιλούμε για κράτη τα οποία βρίσκονται ενώπιον ε, ε, ενώπιον του φάσματος της πτώχευσης, της πτώχευσης της κρατικής. Το να τα βοηθήσουμε δεν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 δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τόσο μικρά, μικρού βεληνικούς, μικρής εμβέλειας ε, μέτρα. Πρόκειται μόνο για πλασέμπο και για τίποτε άλλο. Λειτουργικά προγράμματα λοιπόν τα οποία ήδη δεν μπορεί να, να εξυπηρετήσει η Ελλάδα, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνο τη η Ελλάδα και που καλούμεθα να συγχρηματοδοτήσουμε εμείς προκειμένου να, τα βοηθήσουμε, να, σταθούν, να τη βοηθήσουμε να σταθεί στα πόδια της, δεν ε, είναι λύση. Πρόκειται για μια σοσιαλιστική προσέγγιση την οποία εμείς δεν δεχόμαστε. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν ε, ε, δυνατότητες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που θα μπορέσει να εξασφαλίσει μόνο από το δικό της νόμισμα για να μπορέσει να σταθεί στις ε, διεθνείς αγορές. Αυτό ακριβώς είναι που δεν γίνεται και γι' αυτό ακριβώς αυτή η πολιτική είναι σφαλμένη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για 1,5 λεπτό, ο κύριος Μάτουλα η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση συνεχίζει να μένεται και επηρεάζει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα πολλών κρατών καθώς και την πρόσβασή του στη χρηματοδότηση. Η πρόταση που συζητούμε έχει ως στόχο να επιτύχει συνέργεια μεταξύ δανείων και κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς κράτη-μέλη, τα οποία ούτως ή άλλως λαμβάνουν βοήθεια από, από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ρουμανία. Πρόκειται για έργα τα οποία έχουν έσοδα όπως ε, οι αυτοκινητόδρομοι με διόδια. Στόχο είναι να υποστηρίξουμε παραγωγικές επενδύσεις για τις οποίες υπάρχει ανώτατο όριο συγχρηματοδότηση και κρατική επιχορήγηση. Η κατάσταση είναι εξαιρετική. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε αυτό το σύγχρονο εργαλείο για να επιμεριστούν οι κίνδυνοι μεταξύ ΕΤΕΠ αλλά και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για να τονώσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις και να αρθούν τα εμπόδια στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Η λειτουργία του σχετικού μηχανισμού θα αποτελέσει πρόοδο για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνεχής, το οποίο δεν θα μπορούσε να πετύχει τη μέγιστη απορρόφηση μέχρι την εκπνοή της περίοδου 2013. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Για ένα μισή λεπτό τώρα, το λόγο έχει ο κύριος Σταυρακάκης. Ε, President, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Δανούτα Χούμπνερ για τη μεθοδική δουλειά και την εξαιρετική έκθεσή της όπω και τη συνάδελφο μόιτσα κλέβα για την πολύ καλή έκθεσή τη. δεν θα αναφερθώ στα επιμέρου στοιχεία τη έκθεση μια και οι προηγούμενοι συνάδελφοι τα ανέλησαν διεξοδικά. θα ήθελα όμω να τονίσω ότι με τι προτινόμενε αλλαγέ η πολιτική συνοχή συνεισφέρει ακόμα μία φορά τα μέγιστα στην προσπάθεια ανάκαμψη τη οικονομία την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία δεκάδε χιλιάδε νέε θέσει εργασία αναμένονται να δημιουργηθούν μόνο στην ελλάδα ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί και η ολοκλήρωση του ελληνικού τμήματος των έργων του άξονα 7 του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Φυσικά για να ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία έχουν σταματήσει στις χώρες που θα πλήττονται από την κρίση και να γίνει η όσο δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των συγκεκριμένων μέσων, η μόχλευση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο ή και τρει φορέ μεγαλύτερη από το ποσό που θα δεσμευτεί από τα κονδύλια πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό τώρα το λόγο έχει ο κύριος Χρυσόγελος. Ένα τέτοιο εργαλείο διάχυση του κινδύνου είναι σίγουρα σωστό αρκεί να στοχεύει στην, ε, στην αλλαγή προς κατευθύνσεις που κάνουν την οικονομία πιο βιώσιμη και πιο συμβατή με τους οικολογικούς στόχους γι' αυτό ω ομάδα των πράσινων είχαμε προτείνει το εργαλείο αυτό να βοηθήσει την ενίσχυση επενδύσεων σε τομεί, όπω είναι το τρένο το μετρό εξοικονόμηση ενέργεια και ανανεώσιμε πηγές ενέργεια. φαίνεται όμω ότι ο συμβιβασμό μεταξύ κομισιόν ελληνική κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων οδηγεί σε μια άλλη συμφωνία και σε κάθε περίπτωση θα αφορά ε, ουσιαστικά την ολοκλήρωση έργων αυτοκινητοδρόμων που δεν είναι και οικονομικά βιώσιμη αλλά δεν είναι και οικολογικά αναγκαία σήμερα. όταν ε, υπάρχει μεγάλη κρίση ε, δημοσιονομική έχει μειωθεί η κίνηση των αυτοκινήτων και πολλοί οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι αυτά τα έργα δεν είναι πια οικονομικά βιώσιμα. αν δεν κάνω λάθος και η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων έχει αναφέρει κάτι τέτοιο εμεί λοιπόν θα θέλαμε αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί προ την κατεύθυνση τη πράσινη οικονομία όταν το πρωί ο επίτροπο είπε ότι έχει τεράστιε δυνατότητε η πράσινη οικονομία να δημιουργηθούν είκοσι εκατομμύρια θέσει εργασία στην ευρώπη. γιατί όχι και στην ελλάδα τέτοιε θέσει εργασία με τη χρήση και τέτοιου εργαλείου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Χιούμπνερ για την έκθεση και για την δουλειά που έκανε. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που αιτιολογεί τέτοιες μεθόδους ε, κατ' εξαίρεση. Είναι άνευ προηγουμένου η χρηματοπιστωτική κρίση και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα της κρίσης που γίνονται αίσθητα σε ολόκληρη την οικονομία και την αγορά σε όλη την Ευρώπη. Αν δούμε τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε τώρα, θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ε, τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής να χρησιμοποιηθούν με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο για να ενισχυθούν οι οικονομίες. Και θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Κομισιόν που κάνει την πρόταση αυτή για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας ε, των μέτρων συνοχής και που θα ενθαρρύνει τους ε, ιδιώτες επενδυτές ε, να συμβάλλουν στην χρηματοδότηση των μέτρων αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επιτύχουν τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ελπίζω ότι τα μέτρα αυτά που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση στα κράτη-μέλη ε, θα υλοποιηθούν όντως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα μισή λεπτό, ο κύριος Τσέλερ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν μπορεί να εμποδιστεί βέβαια με την τωρινή πρόταση, ούτε και θα έπρεπε ε, πτώχευση κράτους ε, με την πρόταση για τον του κινδύνου, αλλά μπορούν να, δοθούν, να δοθούν κάποιες λύσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων. Η δημοσιονομική κρίση, η κρίση χρέους ορισμένων κρατών οδηγεί σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση σε εξαιρετικά μέτρα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής συνοχής. Υπάρχουν έργα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν διότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση από τις τράπεζες και γιατί δεν διαθέτουν κονδύλια οι ιδιώτες επενδυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει η πρόταση αυτή να εξασφαλίσει με τον επιμεσμό του κινδύνου περισσότερη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής ε, συνοχής, της πολιτικής, οι οποίες διατίθενται στα κράτη εκείνα τα οποία θέλουν να ε, αξιοποιήσουν αυτά τα μέτρα. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προ την κυρία Χιούπνερ, η οποία διευκρινίζει με τι τροπολογίε τη σημαντικά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την καθιστά πιο σαφή και ξεκαθαρίζει το πώς μπορεί ένα κράτος να ζητήσει την ε, ενεργοποίηση αυτού του μέσου επιμερισμού του κινδύνου. Θα θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση και περίοδο να χρησιμοποιηθεί το, το μέσον αυτόν και να μην προδικάσει τις περαιτέρω εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Σάντσε Σμιτ για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Monsieur le Président. Chers collègues. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ο τεχνικός χαρακτήρας της έκθεσης δεν πρέπει να μας αποτρέψει να την ψηφίσουμε. Ζούμε κρίση, έλλειψη ρευστότητα. Η Ελλάδα ασφυξιά μεταξύ των ημιτελών έργων. Τα έργα αυτά είναι απολύτω απαραίτητα για την οικονομική ανάπτυξη και για την επιστροφή στον δρόμο τη ανάπτυξη. Η Ελλάδα πληρώνει βαρύ τίμημα εκκρεμούν χρέη μισού δισεκατομμυρίου από τους παραχωρησιούχους και κινδυνεύει να πληρώσει περισσότερα λόγω μη τήρησης διαφορών οδηγιών σε σχέση με το περιβάλλον. Έχει κονδυλία η Ελλάδα τα οποία δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει από τα διαρθρωτικά ταμεία. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε την απορρόφηση, κυρίω αυξάνοντα κατά 10% το ανώτερο όριο χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση είναι παράδοξη. Έχουμε κονδύλια και τα οποία δεν μπορούμε να δαπανίσουμε. Επιπλέον, οι χώρες οι οποίες κινδυνεύουν, κινδυνεύουν να πληρώσουν επιπλέον πρόστιμα. Κύριε Χιούμπνερ, κατάφερε να πείσει το Συμβούλιο να δεχθεί την πρόταση της Κομισιόν για να χρησιμοποιηθούν ακριβώς τα διαθροτικά ταμεία ως ταμεία εγγύησης για να υλοποιηθούν επιτέλους αυτά τα έργα με τη συνδρομή των ιδιωτών χρηματοδοτών. Υποστηρίζω την έκθεση αυτή, αλλά θα έλεγα και κάτι περισσότερο. Μας κατηγορούν αδίκως ότι είμαστε ένα εργαλείο επιβολής λιτότητας. Όχι. Αν χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, θα τονώσουμε την ανάπτυξη και θα βελτιώσουμε τα δημόσια οικονομικά στις χώρες που πλήττονται περισσότερο μέσω της υλοποίησης αυτών των έργων για το μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Για ένα μισή λεπτό τώρα, κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση έχει πλήξει τη, τα δημοσιονομικά των κρατών μελών και τις αποταμιεύσεις ε, στις τράπεζες. Αυτό το πρόβλημα ρευστότητας σημαίνει περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για μεγάλη κλιμακό έργα υποδομών και επίση έχει επηρεάσει την εκτέλεση των έργων του Ταμείου Συνοχής. Υποστηρίζω την Κομισιόν σχετικά με τη δημιουργία αυτού του μέσου ευημερισμού του κινδύνου γιατί μπορεί να αποτελέσει ένα καταλήτη για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση ε, για τα έργα αυτά. Πρέπει όμω να υπογραμμίσω ότι οι υπάρχουσε δυσκολίε, δεν επηρεάζουν μόνο τι έξι χώρε, τι χώρε για τι οποίε ε, υπάρχουν ε, σχέσει σχέδια ε, Και ε, υπάρχουν ε, χώρες που εφαρμόζουν μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και δεν έχουν ε, πρόσβαση στο μέσο αυτό. Αν περιορίσουμε λοιπόν ε, την πρόσβαση στο μέσο αυτό μόνο σε ορισμένες χώρες ε, θα στείλουμε ένα λανθασμένο μήνυμα διότι το πρόβλημα ρευστότητας αφορά τους πάντες. Καλό λοιπόν την Κομισιόν να εξασφαλίσει πρόσβαση στο μέσο αυτό για όλες τις χώρες που θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό θα εξασφαλίσει καλύτερη υλοποίηση των έργων και ανάπτυξη και απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα μισή λεπτό τώρα η κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση που συζητούμε απόψε και η πρόταση της ευρωπαϊκής επιτροπής αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια μια έξυπνη απάντηση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης κυρίως για χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα και δρυμύτατα όπως είναι η χώρα μου η ελλάδα. χαιρετίζω λοιπόν ιδιαίτερα θετικά την παρούσα πρόταση για τη δημιουργία αυτού του εργαλείου του μέσου καταμερισμού κινδύνου που δίνει τη δυνατότητα σε χώρες να μπορούν να αξιοποιήσουν τους κοινοτικούς πόρους και να ε, μπορούν να εκταμιεύσουν κεφάλαια από την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων ή άλλο οργανισμό για τη χρηματοδότηση έργων που εκτελούνται με συνεισφορές των διαφορετικών ταμείων και του ταμείου συνοχής. δίνει τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να συμμετέχει ε, στην ε, ε, παραγωγή πλούτου δημιουργία θέσεων απασχόλησης και επαναλαμβάνω για χώρες που υφίστανται ισχυρές περικοπές δημοσίων επενδύσεων όπως είναι η ελλάδα. η ελλάδα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον μηχανισμό αυτό κυρίως για την παραχώρηση αυτοκινητοδρόμων και πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για την επανεκκίνηση της ε, οικονομίας που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μου για να μπει σε μια τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Και τώρα πέραμε στη δικασία Καρστιάη. Τέσσερις συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Ο κύριος Λούχαν, ο κύριος Πάσκα, ο κύριος Φερέιρα και η κυρία Παζέσκου. Ο κύριος Λούχαν για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι συνθήκες στον ιδρύκο τομέα είχαν ως αποτέλεσμα σε ορισμένα κρατημέλη κάποια έργα να μην υλοποιηθούν ποτέ. Πρόκειται για έργα υποδομής, τα οποία θίγονται κατά κύριο λόγο. Οι αναλύσεις δείχνουν ότι οι πόροι για την περίοδο 2010-2013 ανέρχονται σε πάνω από 1.100 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρειαζόμαστε ένα αποδοτικό δίκτυο μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί πολύτιμο πόρο. Και εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο πόρο. Ιδιωτικού πόρου, καθώ και δημόσια κονδύλια. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λύση για όλα αυτά τα προβλήματα. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πραγματικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Με τη σύνδρομη τη ΕΤΕΠ και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Τα έργα αυτά με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν με τη συνδρομή βεβαίω των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου συνοχής. Ευχαριστώ. Ο Πάσκα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερα στην προσπάθεια της Κομισιόν να βοηθήσει ε, στην αντιμετώπιση της κρίσης με τη χρήση καινοτόμων μηχανισμών για τις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες δημοσιονομικής σταθερότητας πολλές ε, ε, επενδύσεις στις οποίες διστάζει να συμμετάσχει ο ιδιωτικός τομέας ε, μπορούν να πραγματοποιηθούν με την διάχυση του κινδύνου μέσω του εργαλείου αυτού που προτείνει η Κομισιόν. Και η χρήση αυτού του μέτρου αιτιολογείται από την κατάσταση του χρέους αυτών των χωρών. Και ο κύριος Επίτροπος δέχτηκε ότι υπάρχουν ε, και κάποιοι ε, κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που ε, εμπλέκονται εδώ. Ε, πρέπει να πω ότι έχω κάποιες ε, αμφιβολίες ε, σχετικά με την σκοπιμότητα αυτών των έργων, διότι αν είναι πραγματικά ε, αποδοτικά αυτά τα έργα και κερδοφόρα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και πρόβλημα συμμετοχής των επενδυτών. Φοβάμαι ότι το μέτρο αυτό δημιουργεί επιπλέον προβλήματα για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Comissão ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ακόμα μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ε, δυσκολιών που ε, αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη-μέλη. Πρόκειται για την χρήση ενισχύσεων χρηματοδοτικών που έχουν ήδη εγκριθεί για τα κράτη-μέλη. Τα ποσά αυτά θα αφαιρεθούν από τα κράτη-μέλη που τα χρειάζονται και θα χρησιμοποιηθούν για να ε, αντισταθμιστούν κάποιες δυσκολίες που δημιουργεί η οικονομική κρίση ε, σχετικά με την ε, εξέβρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης για τα έργα αυτά. Αυτό είναι παράλογο αντί να ενισχυθούν τα κράτη-μέλη που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια, αυτό που γίνεται τώρα είναι ε, ότι προτείνεται ένα μέτρο που θα επιδεινώσει την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Αν κοιτάξετε τα επιτόκια που χρησιμοποιούνται ε, για τα... ή αν δείτε την κατάσταση της Ρουμανίας ή της ε, Πορτογαλίας, δεν είναι σε θέση να απορροφήσουν την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια, κυρία Βαζέσκου. Για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλωσορίζω το συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων δανεισμού και των, ε, της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοπιστωτική σταθερότητας. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η συνέχιση των χρηματοπιστωτικών ε, των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από το ΦΕΝΤΕΡ, από το Ταμείο Συνοχή, σε μια περίοδο πολύ μεγάλης δημοσιονομικής ε, στενότητας. Οι συνέπειε, πιστεύω στι οικονομίε οικονομίες των κρατών που επηρεάζονται από την κρίση θα είναι πολύ σημαντικές και ορατές και μπορούν να οδηγήσουν ε, σε αντιμετώπιση της έλλειψης επενδύσεων που προξένει αυτή η κρίση. Η Ρουμανία γνωρίζει επίσης σημαντικές ε, οικονομικές δυσκολίες που επηρεάζουν την ε, υλοποίηση έργων υποδομής και έτσι οι ε, σημερινέ συζητήσει είναι ευπρόσδεκτε. Το Διεθνέ Ορματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον έχουν συστήσει στην, στην Ρουμανία να αξιοποιήσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματο Ανάπτυξη ω το περισσότερα κονδύλια ευρωπαϊκά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε, και τώρα εκ μέρου Ευρωπαϊκή ο Σεμέτα έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τις παρατηρήσεις τους. Διπιστώνω ότι όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε τις πλέον απειλούμενες χώρες. Το θέμα συζητήθηκε σε διάφορες επιτροπές αλλά και σήμερα στην Ολομέλεια. Θέλαμε με την ευκαιρία να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για εξαιρετικό μέτρο, για μια εξαιρετική κρίση. Δικαιολογείται λόγω της σοβαρής κατάστασης στην Ελλάδα, αν και ορισμένα χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης απαντώνται και αλλούς άλλες χώρες με παρόμοια προβλήματα. Σε εποχή δημοσιονομικών περιορισμών, το να επεκτείνουμε την εφαρμογή του μέτρου σε όλες τις χώρες θα έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Τώρα όσον αφορά το αντικείμενο του νομοθετικού μέτρου. Η πρόταση της Κομισιόν αφορούσε μόνο τα έργα τα οποία εντάσσονται στα εθνικά πλαίσια στρατηγικής. Συμφωνήθηκε στην συνέχεια να διευρύνουμε το πεδίο και εκτός τέτοιων έργων βασιτήσεως του κράτους μέλους και βάση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή. Πιστεύουμε ότι η τελική συμβαστική λύση είναι καλή, διότι λαμβάνει υπόψη και έργα τα οποία εντάσσονται ακριβώ στην πολιτική και τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Εκτιμούμε ότι ένας σημαντικός αριθμός έργων θα φορούν το περιβάλλον μεταξύ αυτών στον τομέα των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ την προσοχή σας στο ότι έργα τα οποία δεν εντάσσονται στην ε, συνοχή ε, θα αντιμετωπιστούν μεγάλη επιφύλαξη. Πρόκειται λοιπόν για έκτακτο μηχανισμό ο οποίος αφορά συγκεκριμένα κρατημέλη. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μηχανισμός διευκόλυνσης ως ένας ε, μηχανισμός ευκαιρίας για να εκμεταλλευτούμε τα διευθυντικά ταμεία. Η πολιτική συνοχή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι μόνο η επένδυση στρατηγική σημασία, αλλά ότι μπορεί να παράσει και βραχυπρόθεσμη βοήθεια εκεί που χρειάζεται. Καλό λοιπόν του βουλευτέ να υποστηρίξουν την νομοθετική αυτή πρόταση. Ευχαριστώ για δύο λεπτά η κυρία Χιούπνερ για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Είναι σαφέ, πιστεύω, από τη συζήτηση και από τα όσα ακούσαμε και από τον Επίτροπο ε, ότι θα χρειαστεί καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων ε, που θα υλοποιήσουν τον κανονισμό αυτών και των κρατών μελών ε, που εμπλέκονται. Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι για κράτη όπως η Ελλάδα θα δοθεί η δυνατότητα για ανάληψη ή επανάληψη μέτρων που έχουν διακοπεί λόγω της οικονομικής κρίσης και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το χειρότερο δυνατό τις σχετικές ρυθμίσεις. Επίσης, Ω εισηγήτρια θα ήθελα να δώσω μια εκτίμηση. Θα ήθελα να πω ότι είχαμε πολύ καλό και επικοδομητικό διάλογο με του και οδησηγητέ αλλά και του ε, συναδέλφου που είχαν την αρμοδιότητα και σύνταξη γνωμοδοτήσεων εκ μέρου των λοιπόν συναρμόδιων επιτροπών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να του ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία συνάδελφε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το θέμα αυτό τη ημερησία διάταξη και Αύριο στις 12 θα γίνει η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην συνεδρίαση, για την πειθαρχία που επιδείξατε και για την ε, αυτοθυσία ως προς την ε, ε, παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξάγεται ε, τώρα ή σε λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, Σερμινής, λέει ο